Is there any chance of starting, Chairman? It is already 10 minutes late. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, Πρόεδρε, ήδη έχουν περάσει 10 λεπτά. Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Άτκινς. Συνήθως, φταίμε μόνο, συνήθως μόνο εμείς ερχόμαστε στην ώρα μας, συνήθως. Bene, allora diamo in... Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας για να σεβαστούμε την ακρίβεια των ε, ήδη και να μην ε, και να φανούμε αυστηροί προς αυτούς που έχουν καθυστερήσει. Έχουμε μπροστά μας ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον, ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μυροσλάβ Λάιτσακ, διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, υπεύθυνο για τις σχέσεις μας με τη Ρωσία, τις ανατολικές γενοτικές χώρες και τα Δυτικά Βαλκάνια. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τις ε, τελευταίες εβδομάδες η περιοχή αυτή ε, διήλθε μια σημαντική κρίση στο Κωσυφοπαίδιο. Ο νεοεκλεγής πρόεδρος υπό ε, υποβλήθηκε σε μια διαδικασία αντισυνταγματικότητας όσο αφορά την εκλογή του. Στην Μακεδονία ε, εκλογές ε, προετοιμάζονται για τις αρχές Ιουνίου. Ε, ως επακόλουθο μια σημαντικής πολιτικής κρίσης, η αντιπολίτευση αποφάσισε να φύγει από, από το Κοινοβούλιο. Στη Βοσνία Ερζεγοβίνη εξακολουθεί να επικρατεί τέλμα δεν υπάρχει ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Μετά από τις εκλογές δεν συγκροτήθηκαν σε σώμα ακόμα οι κυβερνήσεις των πολιτιών. Από ό,τι φαίνεται η χώρα αυτή ε, διέρχεται μια κρίσιμη κατάσταση παρότι βρίσκεται καθοδόν προς την ένταξη στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλβανία τώρα, κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να στείλει επιτόπου μια αντιπροσωπεία, μια αντιπροσωπεία ad hoc για να παρακολουθήσει τις ε, ε, τοπικές εκλογές, τις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση που πρόκειται να δεξαχθούν ως ονούπο. Ε, νομίζω ότι οι δημοκρατικές διαδικασίες στην ε, Αλβανία υπολείπονται πολύ ακόμη. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία να γνωρίσουμε τους γειτονές μας ε, να, να, και να ασκήσουμε κάθε επιρροή που μπορούμε για να συνεργαστούμε για τον εκδημοκρατισμό στην περιοχή. Ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε ένα αυστηρό πρόγραμμα γιατί στις 10 πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία της ψηφοφορίας. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο στον κύριο Μυροσλάβ Λάιτσακ και αναμένουμε με ενδιαφέρον να τον ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι πολύ που έχω την ευκαιρία να σας μιλήσω σήμερα για τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανιών. Μόλις επέστρεψα μάλιστα από την περιοχή. Ο πρόεδρος Μπαρόσο επισκέφθηκε τέσσερις ε, χώρες της περιοχής. Ε, με ενημέρωσε ο Επίτροπος Φίλερ για την ε, επίσκεψη αυτή και θα μπορέσω να μιλήσω για την κάθε χώρα ξεχωριστά. Ξέρω πόσο ενδιαφέρεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την περιοχή και πόσο θέλει να στείλει ένα συνακτικό ενιαίο ευρωπαϊκό μήνυμα. Και στο πλαίσιο αυτό θέλω κι εγώ να έχω έναν υποδομητικό διάλογο μαζί σας. Σερβία, Κωσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο, Βοσία, Ερζεγοβίνη είναι χώρες ε, που θα επισκεφθούμε πριν από τις ε, θερινές διακοπές και είναι μια ευκαιρία να στείλουμε το σωστό μήνυμα. Παρόλε τι προόδου που έχουν σημειωθεί, παραμένουν πολλέ προκλήσει στην περιοχή αυτή. Εκλογέ τοπική αυτοδιοίκηση στην Αλβανία τον επόμενο μήνα, ε, γενικέ εκλογέ στη Σερβία και στο Μαυροβούνιο και επίση στην ε, Κροατία ε, το επόμενο έτος. Η περιφερειακή συνεργασία στα Βαλκάνια συνεχίζεται, έχουν υπογραφεί διμερείς συμφωνίες, πλησιάζει μια σημαντική συνάντηση, η Σύνοδος Κορυφής τον Ιούνιο και υπάρχει μια σημαντική διαδικασία συμφιλίωσης. Αυτό ξεκίνησε την 1η Απριλίου στο Μαυροβούνιο, την Κροατία και το Κωσυφοπαίδιο με εξαίρεση τον Βορρά, αλλά όχι στι υπόλοιπε περιοχέ των Δυτικών Βαλκανίων. Τώρα η κατάσταση στην κάθε μία χώρα ξεχωριστά. Μας ανησυχεί πολύ η πολιτική κατάσταση στη Βοσνία Ερζεβοβίνη. Η κυβέρνηση που σχηματίστηκε τον Οκτώβριο βρίσκεται σε τέλμα. Μια χωρα ξεχωριστα μα ανησυχει πολυ η πολιτικη κατασταση στη βοσνια ερζεβοβινη η κυβερνηση που σχηματιστηκε τον οκτωβριο βρισκεται σε τελμα μια πολιτικη κρίση εξελίσσεται. Η νέα ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν συμπεριέλαβε τα δύο κυριότερα πολιτικά κόμματα της Κροατίας και αυτό δεν είναι καλό. Ταυτόχρονα ο πρόεδρος Ντοβίνκο της ε, Δημοκρατίας της Σέρψκα ε, έχει γίνει στόχος ε, ποινική δίωξης από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα η χώρα κινδυνεύει να χάσει ακόμα περισσότερο χώρο και να μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει επικεντρωμένη στην κατάσταση στη Βοσνία Ερζεγοβένη. Τις ερχόμενες εβδομάδες θα ενισχύσουμε την πολιτική μας παρουσία εκεί με έναν ενιαίο εκπρόσωπο αυτή τη στιγμή αναζητούμε τους αρχηγούς των αντιπροσωπιών που με ισχυρή εντολή και με πόρους στη διάθεσή τους θα, θα πάνε εκεί να παρακολουθήσουν την κατάσταση. Λαμβάνουμε αυτά τα μέτρα σε στενή συνεργασία με τους κύριους εταίρους μας στη διεθνή κοινότητα. Στην Πρίστινα υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχει ένας νέος πρόεδρος, υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις μπροστά τους και πρέπει να τους βοηθήσουμε. Το πιο σημαντικό από απόψη σταθερότητα είναι ο διάλογο. Το περασμένο μήνα ξεκίνησε επιτέλου ο διάλογο. Ο στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να διευκολύνει και να επιτευχθεί πρόοδο στο δρόμο προ την ένταξη και για τι δύο χώρε για να βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων. Ε, η πρώτη συνάντηση ε, έλαβε χώρα το Μάρτιο σε επικοδομητική ατμόσφαιρα και θα ακολουθήσει δεύτερη συνάντηση μετά το Πάσχα. Δεν υπάρχουν θεαματικά αποτελέσματα ακόμη, αλλά πολλές συζητήσεις για πολλά θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των ανθρώπων και κάποια θετική πρόοδος επιτεύχθη ήδη ε, όσο αφορά τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα και την συνεργασία στην περιοχή. Το περιβάλλον είναι δύσκολο. Εμείς παραμένουμε δεσμευμένοι στον διάλογο και το θεωρούμε προτεραιότητα για την περιοχή. Μιλήσαμε για την Αλβανία πολλές φορές. Η κυρία Άστον έστειλε ένα σαφές μήνυμα στην 31 Μαρτίου ε, προς υποστήριξη της αναβίωσης του διαλόγου. Η απουσία άμεσου πολιτικού διαλόγου μεταξύ των κυριότερων πολιτικών δυνάμεων είναι πηγή ανησυχίας και εμποδίζει την πρόοδο το Φεβρουάριο η Ελομέλεια του ε, Κοινοβουλίου εξέτασε την κατάσταση στην χώρα αυτή και κατά την επίσκεψη των σχετικών εκπροσώπων στα Τύρανα τονίστηκε η ανάγκη επανέναρξης του διαλόγου. Στις 28 Μαρτίου πήγα για τρίτη φορά στη χώρα μετά από τον τέλος του Γενάρη και τόνισα το σημείο αυτό. Συνεργαζόμαστε και με τους διεθνείς εταίρους μας, τις Ηνωμένε Πολιτείες, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ε, θε, μια κάναμε μια συνάντηση στο τοπικό κοινοβούλιο και ήρθαμε σε επαφή με πάρα πολλούς εκπροσώπους των περισσότερων πολιτικών κομμάτων. Ε, σας ενθαρρύνω ε, να εκφράσετε συλλογικά την πλήρη υποστήριξή σας προς όλες αυτές τις προσπάθειες, τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς την αντιπολίτευση, να γεφυρωθούν οι υφιστάμενες ε, ε, διαφορές και να μπορέσουν να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πλαίσιο για τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το διακύβευμα στην ε, Αλβανία είναι πολιτικά και συμβολικά πολύ υψηλό. Ε, πάντως μια έκκληση για διάλογο έχει τη χρησιμότητά σας. Ε, τώρα για την πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας οι εξωτερικές υπηρεσίες κατέγραψαν την έκθεσή σας για τη χώρα αυτή που υιοθετήθηκε τον Απρίλιο και την έκκληση για συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Δώσατε την έμφαση στις καλές γειτονικές σχέσεις, σχέσεις καλής γειτνίασης σημαντικό για όλες τις χώρες. Γενικά η πολιτική κατάσταση κυριαρχείται από τις επερχόμενες εκλογές. Μπορεί να υπάρξει απώλεια χρόνου όσο αφορά την ε, ατζέντα των ε, μεταρρυθμίσεων που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα αυτή. Ενθαρρύνουμε τόσο τη σημερινή, ε, το σημερινό συνασπισμό όσο και την αντιπολίτευση να διεξαχθούν ομαλά οι εκλογές Τέλος, στηρίζω τις προσπάθειες όλων των πλευρών για ελεύθερες, δίκαιες, διαφανείς και δημοκρατικές εκλογές. Αυτό είναι το μέλλον που απέστειλε την περασμένη εβδομάδα και ο πρόεδρος Βαρόσο. Έχουμε μια νέα κυβέρνηση στο Βελιγράδι. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Πρέπει να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις το 2011 θα υπάρξει ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει μεγάλη σημασία στη χώρα αυτή και θα υπάρξουν πολλές προσπάθειες ιδίως για το βόρειο κοσυφοπέδιο. Ε, η επίλυση του ζητήματος του κοσυφοπεδίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για το ευρωπαϊκό μέλλον της ε, Σερβίας. Οι σχέσεις μας με το Μαυροβούνιο είναι σταθερές, έχουν παγιωθεί. Ε, τον Ιούνιο θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Συμβουλίου Ένταξης και θα εξεταστούν οι σχετικές προτεραιότητες. Η γνώμη της Επιτροπής θα αποτελέσει βάση για το μέλλον. Το Μαυροβούνιο πρέπει να παρέχει ε, σταθερότητα. Είναι μια χώρα που έχει καλές ε, σχέσεις γειτνίας με τις γειτονικές χώρες. Βέβαια, σε σχέση με τη Σερβία υπάρχουν κάποιες εντάσεις. Οι καλές σχέσεις γειτονίας είναι μια αρχή στην οποία εκφράζουν τη δέσμευσή τους και οι δύο πλευρές. Η Κροατία βρίσκεται σε κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων. Στις 19 Απριλίου εδώ στις Βρυξέλλες θα υπάρξει μια συνάντηση και αναμένουμε πολλά από αυτήν. Το πιο ευαίσθητο σημείο είναι η δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη δικαιώματα. η έκκληση του... στο Ζάγκρεπ την περασμένη εβδομάδα ανακουφίστηκα με την έκκληση συνέχισης προσπαθειών που απέφθηνε στους, προε... στους πρωθυπουργούς των δύο κρατικών οντοτήτων ο πρόεδρος της χώρας. Κυρίες και κύριοι, η εικόνα των Δυτικών Βαλκανίων είναι περίπλοκη. Η κάθε χώρα έχει τις δικές της προκλήσεις να αντιμετωπίσει μένα, αλλά όλες μοιράζονται κάτι κοινό, την ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία τις βοηθάει να ε, εφαρμόσουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις και να φέρουν το οικονομικοπολιτικό τους σύστημα πιο κοντά στο ευρωπαϊκό. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι χώρες αυτές θα εξακολουθήσουν να επιδιώκουν την ευρωπαϊκή ατζέντα και να παρέχουμε τη σχετική υποστήριξη προς αυτές. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, δόκτωρα Λάιτσακ. Έχουμε μια ομάδα συναδέλφων που ζήτησαν να παρέμβουν. Ε, θα τους δώσω τρία λεπτά στον καθένα, έτσι ώστε όλοι να μπορέσουν να εκφράσουν τη γνώμη τους και θα δώσω το λόγο στην επικεφαλής της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις μας με, την Ανατολ... με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, τον κύριο Κούκατ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μας περισσεύουν τα τρία λεπτά. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λάιτσακ για την παρουσία του εδώ. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις ε, δραστηριότητες του στην περιοχή αυτή. Είναι μια περιοχή που απαιτεί μια συνεχή ενασχόληση. Νομίζω ότι κάλυψε όλα τα ουσιώδη θέματα που έχουν να κάνουν με την κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια και ανεφέρθηκε στο πρακτέον για το άμεσο μέλλον. Εγώ θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα αυτό το οποίο ανέφερε, ότι δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή προσέγγιση να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση στη Δυτικά Βαλκάνια μαζί με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Κομισιόν. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς ιδιαίτερα είναι η συνδιάσκεψη για τα Δυτικά Βαλκάνια που θα περιλαμβάνει και πολλούς ομιλητές από τα Δυτικά Βαλκάνια και ο στόχος μας είναι να υπογραμμίσουμε και στη συνδιάσκεψη αυτή το σημείο αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο να τονιστεί. Τώρα, <clears throat> μπορεί να θέσει κανείς μια πλειάδα ερωτήσεων και ο κύριος Λάτσεκ έχει καλύψει όλα τα θέματα περίπου. Θέλω όμως να θέσω τρία ερωτήματα για, θέλω να αναφερθώ σε τρεις χώρες. Η Αλβανία καταρχήν. Έχουμε επενδύσει πάρα πολλά για να βοηθήσουμε την αλβανική πολιτική τάξη να βγει από την κρίση αυτή η οποία οδηγεί σε μια κατάρρευση των προοπτικών της Αλβανίας. Και εάν δεν επιληθεί με πολιτικό τρόπο αυτή η κρίση θα είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για ταχεία πρόοδο της Αλβανίας στο μέλλον. Οι τοπικές εκλογές λοιπόν, οι δημοτικές εκλογές της 8ης Μαΐου, εάν προετοιμαστούν σωστά και αν διεξαχθούν με δημοκρατικό και διάφορο τρόπο, μπορούν να δώσουν ένα θετικό μήνυμα. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν, ποια είναι η άποψή σας κύριε Λάτσεκ, τι μπορεί να γίνει για να μην επαναληφθεί η κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε μετά από τις ε, πρόσφατες βουλευτικές εκλογές που συνεχίζεται ακόμα και τώρα αυτή η έκριθμη κατάσταση. Για την Μακεδονία επίσης αναφερθήκατε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητούσε την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων ένταξης για τη χώρα αυτή. Αλλά εάν δεν επιληθεί το πρόβλημα του ονόματος θα είναι και πάλι να επιτευχθεί οποιαδήποτε πραγματική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τη χώρα αυτή. Θα είναι πολύ σημαντικό η νέα κυβέρνηση που θα προέλθει από τις εκλογές με την φρέσκια εντολή που θα έχει πάρει να προσπαθήσει να προχωρήσει προς την κατεύθυνση μιας λύσης η οποία θα εξασφαλίσει και μια επιτάχυνση της διαδικασίας για την ένταξη της χώρας αυτής στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το Κωσυφοπαίδιο, είπατε ότι στην Πρίστινα βλέπετε πια να υπάρχουν σαφέστερες ε, ε Τι ακριβώς εννοείται εδώ. Ευχαριστώ κύριε Κούκαν. Ο λόγος στην κυρία Πακ, συγγήτρια για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Τρία λεπτά παρακαλώ. Το äh, κάθε επιτυχία στην μελλοντική σας εργασία στο Κοσμοπέδιο, λέει η κυρία Πακ. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα για την ε, Βοσνία, μετά για την Αλβανία και το Κοσμοπέδιο η κατάσταση στη Βοσνία έχει επιδεινωθεί βαθμία. Οι εθνικές διακρίσεις και διχόνοιες είναι ακόμα μεγαλύτερες από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Και φυσικά οι πολιτικοί εκμεταλλεύονται πλήρως στο έπακρο της εθνικιστικές εντάσεις και δεν κάνουν τίποτα για να βοηθήσουν τους ε, ανθρώπους να αποκτήσουν καλύτερες υποδομές, καλύτερη κατάρτιση, να έχουν καλύτερη παροχή ενέργειας και άλλων βασικών πόρων. Νομίζω λοιπόν ότι ο τρόπος με τον τρόπο έγινε ο σχηματισμός αυτής της κυβέρνηση δεν ήταν ο καλύτερος, αλλά εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και μόνο το συνταγματικό δικαστήριο της χώρας μπορεί να επιληθεί ενό τέτοιου θέματο. Είπατε ότι υπάρχει μια ενισχυμένη πολιτική παρουσία. Τι σημαίνει αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο παρούσα. Ποια είναι τα εργαλεία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να επιτύχει να υπάρξει πρόοδο στην περιοχή αυτή. Έχουμε μονάχα το μοχλό της βοήθειας. Λέμε ότι άμα δεν πράξετε το α και το β δεν θα πάρετε το παραμικρό κονδύλιο από εμά. Αλλά αυτό μονάχα έχουμε στα χέρια μας. Είναι κρίμα να χρειαστεί να καταφύγουμε σε τέτοια ε, μέσα, αλλά η εμπειρία μου μου έχει δείξει ότι χωρίς πίεση δεν μπορεί να επιτευχθεί τίποτα και δεν μπορεί να υπάρξει πραγματικά πρόοδος εάν δεν ασκήσει πίεση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το ένα στοιχείο το οποίο ε, ε θέλω να αναφέρω. Χρειαζόμαστε μια νέα συμφωνία του Dayton, μια Dayton Sin. Μήπως θα ήταν δυνατό να πούμε ότι θα πρέπει να προβούμε σε διαπραγματεύσει για μια νέα συμφωνία για την περιοχή αυτή. Και εδώ ούτε η Κομισιόν ούτε το Συμβούλιο έχει αναλάβει σωστά, το, έχει αντιμετωπίσει σωστά αυτό το πρόβλημα. Η Ομοσπονδία αυτή έχει τη μορφή που έχει στη Βοσνία. Δεν φταίνε οι άνθρωποι. Αλλά όπως έχει τώρα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και έχει και αρνητική επίπτωση η λειτουργία της στους γείτονές της. Είναι πραγματικά έσχος ότι δεν έχουμε ακόμα κάποιον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια χώρα που χρειάζεται τόσο κατεπηγόντω να έχει ένα πραγματικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος θα διαδραματίσει τον αντίστοιχο ρόλο. Για το κοσμοπέδιο. γνωρίζω ότι τα πράγματα τα οποία λαμβάνουν χώρα εκεί δεν είναι ιδιαίτερα θετικά. Αυτό το οποίο όμως εμένα με ενοχλεί είναι ότι εμείς είμαστε απόντες. <clears throat> Όχι μόνο εμείς, Υπάρχει ένα κουαρτέτο από το οποίο μόνο οι τρεις είναι παρόντες και εμείς ποτέ είμαστε παρόντες. Και για το θέμα της παρακολούθησης των εκλογών στην Αλβανία, εγώ είχα πει ότι δεν πρέπει να στείλουμε παρατηρητές. Όλες τις προηγούμενες εκλογές τις είχαμε παρακολουθήσει. Είχαμε <clears throat> πριν από αυτές τις εκλογές που έλαβαν χώρα τι ε, προτελευταίε εκλογέ, οι οποίε ήταν πολύ επιτυχεί και είχαμε πει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά οι τελευταίε εκλογέ δεν ανταποκρινόντουσαν στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ευχαριστώ, κύριο Κάτσιν, εισηγητή για τη Σερβία. Τρία λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, πρόεδρε, κύριε Λάιτσακ, καλώ ήλθατε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις προσπάθειες που έχετε κάνει και εσείς και ο πρόεδρος της Επιτροπής και ο Επίτροπος, ο Φίλε, την Παρασκευή να στη Βοσνία Ζεγοβίνη, όπως και εσείς. Δεν θέλω να υποτιμήσω εδώ την κατάσταση που επικρατεί εκεί, αλλά θέλω να υπογραμμίσω ότι είναι πήγον κάτι να προσφέρουμε, γιατί οι ίδιοι δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτε. Οπότε εμείς πρέπει να κάνουμε το μεγάλο βήμα. Η κατάσταση στην Βοσνία φυσικά και είναι δύσκολη, όπως και στην Αλβανία. Όμως αυτό που θέλω εδώ να αναφέρω είναι το θέμα της Μακεδονίας. Έξι χρόνια δεν έχουμε καμία διαφορά, καμία αλλαγή. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κακό παράδειγμα. Αυτό που πραγματικά χρειάζεται λοιπόν είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος όσον αφορά το θέμα του ονόματος. Χωρίς ε, συμβιβασμούς ε, δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα, την αλήθεια ποιος είναι κομμάτι της λύσης και ποιος είναι κομμάτι του προβλήματος. Θέλω να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε αυτοί που είναι το πρόβλημα να αλλάξουν και να αρχίσουν να συμπεριφέρονται κάπως διαφορετικά. Να αλλάξουμε τον χειρότερο εχθρό σε γείτονα, να έχουμε καλές σχέσεις με τους γείτονες και όλοι οι γείτονες μαζί να προσπαθήσουν να βρουν μια διέξοδο. Όσον αφορά το κοσυφοπέδιο τώρα έχω μια πρακτική ερώτηση. Ξέρετε, γνωρίζετε τον καινούριο πρόεδρο κύριε Λάβτσικ, νομίζω ότι κανείς. Και υπάρχει και κάτι άλλο όμως που θέλω να πω εδώ ως εισηγητής για το θέμα της Σερβίας. Είναι πραγματικά περίεργο μετά τις εκλογές στο Κωσιβοπέδιο, οι Σέρβοι αποτελούν μέρος της λύσης. Οι Σέρβοι αποτελούν ε, μέρος της ε, κυβέρνησης στο Κωσιβοπέδιο με τρεις υπουργού, με έναν αναπληρωτή πρωθυπουργό, ο οποίος είναι υπεύθυνο για την τοπική σερβική κυβέρνηση. Έχουν τους δικούς τους δημάρχους, όμως οι δήμαρχοι αυτοί δεν αναγνωρίζονται από το Βελιγράδι. Δεν αγνοούνται πλήρως. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε ένα τρόπο ώστε το Βελιγράδι, αν μη τι άλλο, να τους αφήσει στην ησυχία τους. Να τους επιτρέψει να λειτουργήσουν υπέρ του σεβεκού πληθυσμού στους δήμους τους. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί ανάμεσα στη Σερβία και το Κωσυφοπαίδιο. Προτείνω λοιπόν κύριε Λάιτσεκ να, να συνεχίσουν και οι δύο πλευρές να συμμετέχουν σε μια συζήτηση και αυτό να είναι στην ημερήσια διάταξη ζητάω μια πρακτική λύση για τους δημάρχους ώστε να μπορούν να ασχοληθούν με τους Σέρβους που εξακολουθούν να βρίσκονται στο κοσυφοπαίδιο. Αυτό πρέπει να φροντίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κάτσιν. Ο λόγος στην κυρία Λούνατσεκ, εισηγήτρια για το κοσυφοπαίδιο. Τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και εκ μέρους μου θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λέτσικ που ήρθε εδώ στην Επιτροπή μας. Και εγώ θα επικεντρωθώ στο Κωσυφοπαίδιο. Και θα συνεχίσω μετά από αυτά που είπε ο συνάδελφος Κατσίν πριν από λίγο. Όντως, στις 15 είχαμε μια συνάντηση με κάποιους από τους δημάρχους και τους αναπληρωτές ορισμένων δήμων στο Κωσυφοπαίδιο. Ήρθαν, μας μίλησαν για τα προβλήματά τους και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο προλαλής ότι χρειάζονται την υποστήριξή μας και ότι είναι αναγκαίο για αυτού εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκαθαρίσουμε στο Βελιγράδι ότι πρέπει να του στηρίξουν τους δήμους αυτούς και τους δημάρχους. Και στο Βορρά, όπου εξακολουθούν υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ε, θέλω να σας ρωτήσω για κάτι όμως. Τι πιστεύετε εσείς για αυτό που κάνουμε εμείς Α, όσον αφορά την απογραφή στην ε, περιοχή με τους διάφορους δήμους στο νότο, εντάξει, αλλά στο βορρά υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Παρόλο που υπήρξε συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Σφέκοβιτς, τον ε, Πρωθυπουργό, δεν υπάρχει στήριξη, παρόλο που υποσχέθηκε. Εσείς λοιπόν τι μπορείτε να κάνετε, τι γίνεται από την πλευρά μας ώστε να υπάρξει συμμετοχή στην απογραφή αυτή. Όσον αφορά τώρα το διάλογο ανάμεσα στο Κωσυφοπαίδιο και τη Σερβία. Και εγώ πιστεύω ότι είναι μια σημαντική στιγμή, υπάρχει πρόοδος, κάτι γίνεται. Η προβληματική είναι ότι ο κόσμος στο κοσυφοπαίδιο γενικά δεν πιστεύουν ότι κάτι γίνεται για αυτούς. Εγώ προσπαθώ να τους το πω κι άλλοι προσπαθούν να του το πούν, αλλά η γενική αντίληψη που επικρατεί στον πληθυσμό δεν είναι αυτή. Ε, νομίζουν ότι ο διάλογο είναι για τη Σερβία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό από τη δικιά σα την πλευρά, από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση να φανεί τι έχει να κερδίσει το, το πεδίο. Τα τεχνικά στοιχεία είναι σημαντικά, αλλά πρέπει να γίνει κάποια πρόοδο και όσον αφορά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Τι μπορείτε να μα πείτε λοιπόν πάνω σε αυτό παρακαλώ. Και κάτι άλλο που αναφέρατε εσεί ο ίδιο. Μιλήσατε για τη διαδικασία ε, σύμπτυξης των υπηρεσιών. Όπως είπε και η κυρία Πακ, η αντίληψη που επικρατεί σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διάφορες λειτουργίες, διαφορετικά καθήκοντα, αυτοί όμως πηγούνται τις διαδικασίες, είναι τελικά οι Ηνωμένε Πολιτείε. Έτσι όπως αντιλαμβάνομαι εγώ τα πράγματα, θα υπάρξει μια προσωρινή λύση για το USR και ότι δεν ξέρουμε ακόμα ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα ώστε να εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση από έναν άνθρωπο στην περιοχή. Σε αυτό πρέπει να στοχεύσουν οι προσπάθειές μας, γιατί μας βλέπουν σαν να είμαστε διάφορα θεσμικά όργανα, διάφοροι άνθρωποι και που δεν εκφραζόμαστε με μία φωνή. Ναι, ναι, πρόεδρε, τελειώνω. Ένα πραγματάκι ακόμα για την Κροατία που θέλω να σας ρωτήσω. Ξέρω ότι πήγε και ο κύριος Μπαρόσο και ο κύριος Φίλαν αλλά εγώ φοβάμαι ότι στην Κροατία, πέρα από την πρόοδο που κάνει η κυβέρνηση εκεί, η κοινή γνώμη αναρωτιέται, θέλουμε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς δεν ενθαρρύνουμε αυτή την ε, θέση υπέρ ε, της ένταξης. Εσείς τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει περισσότερο ώστε ο κόσμος να θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λούνατσεκ. Ο λόγος στον κύριο Τάνοκ, εισηγητή για το Μαυροβούνιο. Παρακαλώ τρία λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, διαδικαστικά θα ήθελα να πω κάτι. Τους τελευταίους δύο μήνες η ομάδα μου έχει ίσο αριθμό βουλευτών με τους πράσινους, επομένως θα πρέπει να υπάρχει εναλλαγή μεταξύ μας σε σειρά προτεραιότητα. Ίσως το θέμα αυτό θα πρέπει να το δείτε, γιατί το τελευταίο καιρό δεν πάντα προτεραιότητα στους πράσινους και όχι σε εμά. Ναι, ναι, είναι η δύναμη της συνηθίας, λέει ο κύριος Τάνοκ. Κύριε Λάτσερ, καλώ ήλθατε εξ ονόματο τη ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Ω μόνιμο συζητητή για το Μαυροβούνιο, θέλω να σα χαιρετήσω και εγώ προσωπικά. Μπορείτε να μα δώσετε κάποιο χρονοδιάγραμμα για τι διαδικασίε διαπραγματεύσεων του Μαυροβουνίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπατε ότι είναι στο σωστό δρόμο, <clears throat> αλλά ακόμα οι διαπραγματεύσει δεν είναι γνωστό πότε θα ξεκινήσουν. Μια ημερομηνία θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Επίση, για την Μακεδονία, την πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία. Τι μπορούν να κάνουν τα κάτι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρξει μια λύση, μια συνολική λύση για το όνομα, κάτι το οποίο εμποδίζει μέχρι στιγμή τη διαπραγματεύσεις της Μακεδονίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα γίνουν πρόορε εκλογέ τον ε, Ιούνιο και ίσω αυτό θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα αυτό για να μην το χρησιμοποιήσουν προ όφελό του οι σκληροπυρηνικοί που θέλουν να γυρίσουν την πλάτη του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, επειδή έχει χρονίσει τόσο πολύ το θέμα του ονόματος για το διάλογο κοσφοπεδίου Σερβίας, τι μπορεί να προκύψει σε μορφή πρακτικών ρυθμίσεων από αυτό το διάλογο και γιατί, δεν, γιατί έχει αποκλειστεί εκ των προτέρων οποιαδήποτε σκέψη διχοτόμησης του κοσφοπεδίου ενώ στις διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Παλαιστίνης μια ανταλλαγή γης για ειρήνη θεωρείται ότι είναι η σωστή λύση του προβλήματος. <clears throat> και πάλι για το κοσφοπέδιο. Είχαμε ένα εκπρόσωπο πριν από λίγε μέρες ενώπιον της Επιτροπής μας για, <clears throat> για το λαθρεμπόριο ανθρωπίνων οργάνων και ακούσαμε και εκπροσώπους του, της κυβέρνησης του Κωσυφοπεδίου. Τι ακριβώς κάνετε εσείς για να μελετήσετε, να ερευνήσετε αυτές τις σοβαρές καταγγελίες και πώς θα προστατεύσετε τους μάρτυρες που θα καταθέσουν εάν εμφανιστούν για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Μετά από τους εισηγητές σας περάσουμε στους συντονιστές. Δύο λεπτά. Κύριε Βίγκεν. παρακαλώ. σας ευχαριστώ και εγώ κύριε πρόεδρε. Μία παρατήρηση. Έχουμε την εντύπωση ότι η κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια δεν εξελίσσεται θετικά. Δυστυχώς, μόνο μια ιστορία επιτυχίας υπάρχει αυτή τη στιγμή, είναι το Μαυροβούνιο. Στις άλλες χώρες ή αποτελματώνεται η κατάσταση ή επιδεινώνεται και κινείται ανάστροφα από αυτό το οποίο θέλαμε. Μίλαμε πάντα για τη λεγόμενη κόποση διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά φαίνεται ότι και η ίδια η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων έχει κουραστεί. <clears throat> Γιατί φαίνεται τόσο μακρινή η προοπτική της ε, ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε η πολιτική της περιοχής δεν είναι έτοιμη να θυσιάσουν τη δημοτικότητά τους με μεταρρυθμίσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα οδηγήσουν σε εκλογικές ήττες στη συνέχεια. Επομένως, εστιάζουν την προσοχή τους σε τελείως κοντόφθαρμους στόχους πολλές φορές. <clears throat> Γι' αυτό μαζί με τον κύριο Φιούλε θα πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη επινοητικότητα και να δούμε τι βήματα μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε σε αυτή την ε, ε, χρονική περίοδο τις μεταρρυθμίσεις και την ε, υλοποίησή τους από, την πολιτική, από τις πολιτικές ελίτ της περιοχής αυτής. Έχουμε και εμεί τι ευθύνε μα, αλλά πρέπει να σαφές ότι η ευθύνη είναι κοινή και από τη δική μα πλευρά και από την δική του πλευρά. Για τη Βοσνία. Φαίνεται ότι η πολιτική μας για τη Βοσνία δεν έχει λειτουργήσει, όπως είπε και η κυρία Πακ. Τα πράγματα πηγαίνουν προς το χειρότερο. Εξακολουθούν να υπάρχουν οι αντιπαραθέσεις, ο διχασμός γίνεται πιο βαθύς. Μήπως θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την προσέγγιση μας προς τη Βοσνία. Πάντα είναι πιο εύκολο <clears throat> να επιμένει κανείς στην τωρινή πορεία να ζητάει να ασκήσει πίεση στους Βοσνίους για να ανταποκριθούν. Αν όμω δεν πιστεύουν ότι αυτά τα οποία εμεί προτείνουμε και για τα οποία πιέζουμε αποτελούν τη λύση, δεν θα επιτύχουμε τελικά απολύτω τίποτα. Από την άποψη αυτή σας ρωτώ, είσαστε έτοιμος να αναθεωρήσετε τη σκέψη σας για τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Βιγγένιν. Ε, ένας καινούριο εισηγητής, Κάουντης, εισηγητής για την Αλβανία. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λάιτσεκ για την ενημέρωση που μας έκανε. Ερώτηση πρώτη σχετικά με το κοσυφοπαίδιο. Το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την αντισυνταγματικότητα της εκλογής του, του νέου Προέδρου αποτελεί παράγοντα προφανώς πολιτικής αστάθειας και πώς βλέπετε να αντιμετωπίζετε. Μπορεί να συνεχιστεί η πολιτική ζωή όταν επικρέμαται μια τέτοια α, και ένα τέτοιο συνταγματικό πρόβλημα. Δεύτερο, σε σχέση με την Αλβανία, ε, διαψεύστε με ή επιβεβαιώστε με, τα σημάδια δεν είναι ενθαρρυντικά. Οι εκλογές και η εκλογική καμπάνια δεν είναι άμυροι, ε, χωρίς κρούσματα βίας και είμαι ανήσυχος αν πράγματι θα έχουμε ε, δημοκρατικές και ελληνικές εκλογές. Και το ερώτημα είναι, η δική σας η άποψη ποια είναι και η συμμετοχή και η παρα, παρουσία εκεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης των παρατηρητών πιστεύετε ότι συμβάλλει, εγώ είμαι σύμφωνος, δεν έχω καμία αντίρρηση να πάει εκεί η αντιπροσωπεία, θα συνέβαλε ώστε να έχουμε ομαλή εξέλιξη των πραγμάτων. Και η τελευταία ερώτηση, μια γενικότερη ερώτηση. Κύριε Λάιτσεκ, επισκέπτεστε συχνά την περιοχή, ε, συζητάτε με τις κυβερνήσεις, με τις πολιτικές δυνάμεις. Ποια εικόνα έχετε αποκομίσει. Τι περιμένουν τελικά από εσά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' επέκταση περιμένουν να δώσουμε λύση εμείς σε προβλήματα που δεν μπορούν να λυθούν. Περιμένουν να είμαστε ένας αμερόληπτος διαιτητής στα προβλήματα που έχει η περιοχή ή θεωρούν ότι η δική σας παρουσία εκεί, το δικό μας εν πάση περιπτώσει ενδιαφέρον αποτελεί εξωτερικό παράγοντα που δεν θα τους δώσει ικανοποιητική λύση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Χούντι. Για να δώσουμε χρόνο στον καλεσμένο μας να απαντήσει, οι επόμενες παρεμβάσεις, συγγνώμη, λυπάμαι πολύ για τους συναδέλφους, θα περιοριστούν σε ένα λεπτό. ένα λεπτό. Ďakujem pána do parlamentu a ma, že Ευχαριστώ. Και καλώς ήρθατε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάντα με χαρά σας βλέπουμε, λέει η κυρία Μπρίζατσικ, εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Έχετε μεγάλη εμπειρία όσον αφορά τα Βαλκάνια. Εμένα με ενδιαφέρει το Μαυροβούνι. Και δεν θα ζητήσω κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία γιατί ξέρω ότι δεν είναι δικιά σα ευθύνη. Θα ήθελα όμω να ξέρω ποιε είναι οι προοπτικέ που υπάρχουν όσον αφορά το Μαυροβούνι σήμερα. Πώ εξελίσσεται η κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ιμπρίζετζιτ. Πάρα πολύ σύντομη. Σεβαστήκατε το χρόνο. Μπότσκουρ, ένα λεπτό. Ehm, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όσον αφορά τη Βοσνία, έχω μια ερώτηση. Ποιε ήταν οι πρώτε αντιδράσεις όσον αφορά την στρατηγική για το μέλλον που πρότεινε στι 21 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βοσνία εντυπωσιάστηκε. ποιε είναι οι εντυπωσει τη και ποιες οι αντιδράσεις από την τετραμερή όσον αφορά την στρατηγική αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα λειτουργήσει εξάλλου, κατά τη γνώμη σας λειτουργήσει για τους ανθρώπους. Και η τελευταία μου ερώτηση. Είσαστε ο αντιπρόσωπός μας. Πώς θα λειτουργήσει, γιατί τον τελευταίο καιρό φαίνεται ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, δύσκολη η Ευρώπη μιλάει με μία φωνή. Δεν θα πρέπει να υπάρχει όντω ένα άτομο που να εκφράζει με μία φωνή την Ευρώπη, αντί κάθε χώρα χωριστά να εκπροσωπείται. Ευχαριστώ κυρία Μποσκούρντ. Βάγγελ, για ένα λεπτό. Ε, Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το γεγονός ότι η Βοσνία Ζεγοβίν είναι στη μέση και γεωγραφικά και πολιτικά στη μέση της περιοχής των ε, Δυτικών Βαλκανίων που ασχολείται με αυτήν ο κύριο Λάτσεκ. Έχω ένα πρόβλημα όμως όταν προσπαθούμε σε μία συζήτηση μονάχα όπω και σήμερα να καλύψουμε όλη αυτή την περιοχή. Γιατί η φύση των προβλημάτων σε διαφορετικές χώρες είναι τελείως διαφορετική. Και αν προσπαθούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε συνολικά την περιοχή, πάντα υπάρχει η πίεση τη <clears throat> ομοιομορφία για τη Βοσνία. Δεν πρέπει να εστιάσουμε στο τι έκανε ποιο ή πότε ή τι και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας να βρεθεί κάποιος που να εκπροσωπεί όλο τον κόσμο στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Αυτό είναι ένα πολιτικό πρόβλημα το οποίο μόνο με μια περιφερειακή προσέγγιση μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή χρειάζεται μια υψηλού επίπεδου πολιτική συνδιάσκεψη για να μπορέσει να αποφασιστεί το μέλλον της Βοσνίας αλλά και της Ερζεγοβίνης. Και κλείνω λέγον ότι θα πρέπει να επιτρέψουμε στην Κροατία να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα προς την πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βάγκελ. Κλείνει η συζήτηση. στην Άρου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσετε τις ερωτήσεις μας. Μια παρατήρηση. Όσον αφορά την Αλβανία, αν μη τι άλλο, είναι προφανέ ότι δεν έχουμε καταφέρει να εκφραστούμε με μία φωνή και τα αποτελέσματα είναι από κακά έω πολύ κακά. Εμεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλε οι πολιτικέ ομάδε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέλαμε να υπάρχει αυτή η έκφραση με μία φωνή. Ξέρετε ότι τελευταία άλλαξαν οι κανόνες και ότι με τους νέους κανόνες λέμε έχουμε καταλήξει πρώτα να ψηφίζουμε ένα νόμο και μετά να το συζητάμε. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε την άποψή σας γι' αυτό. Και κάτι τελευταίο, όπως ξέρετε, τελευταίο πρόεδρος του Αλβανικού Κοινοβουλίου με κατηγόρησε για διαφθορά. Είναι απαράδεκτο. Και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου τρεις φορές προσπαθεί να πείσει την πρόεδρο είτε δημόσια να ζητήσει συγγνώμη ή να αποσύρει τις κατηγορίες της, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ευχαριστώ αγαπητέ κύριε Μποστινάρου. 11 ε, παρεμβάσεις. Έχετε 10 λεπτά για να απαντήσετε. Ξέρω, ξέρετε ότι είναι αδύνατο να το κάνετε και γι' αυτό θα τα καταφέρετε παρόλα αυτά να απαντήσετε. Ευχαριστώ, πολύ και ευχαριστώ για τα ερωτήματα που θέσατε. Είναι μεγάλη ευχαριστήση για μένα να είμαι εδώ. Όχι μόνο είμαι υπεύθυνο για τα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και για την ανατολική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ουκρανία, Μολδαβία, Λευκορωσία, Κάφκασος. Για τα ερωτήματά σας λοιπόν. Για τον κύριο Κούκαν, η Αλβανία, τι περαιτέρω μπορούμε να πράξουμε. Νομίζω ότι έχουμε κάνει πολλά για να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση στην Αλβανία μετά από τα τραγικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στο τέλος Ιανουαρίου. Το μήνυμά μας έχει δοθεί με σαφήνεια. Ήμασταν σε θέση να μιλήσουμε με ενιαία φωνή, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μαζί και με τις ΗΠΑ και τον ΟΑΣΕ. Ξεκινήσαμε μία προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά μετά τις εκλογές. Πρέπει να είμαστε συνεκτικοί και να συνεχίσουμε να τονίζουμε την ανάγκη πολιτικού διαλόγου και της επιστροφής στην ομαλότητα της πολιτικής ζωής και επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι πρέπει στο βαθμό του δυνατού όλες αυτές οι εκλογές να γίνουν με αμερόληπτο τρόπο και να αναλυθούν όλα τα απαραίτητα πολιτικά μέτρα για την επιτεύξη αυτού του στόχου. Η πίεση από τη δική μας πλευρά λοιπόν θα πρέπει να είναι παρούσα για να ξέρουν οι Αλβανοί ότι παρακολουθούμε αυτά που κάνουμε και τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθούν οι εκλογές. Για την πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, για το όνομα είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί αμέσως μετά τις εκλογές και τη δημιουργία μιας κυβέρνησης εκεί. Εκεί είναι το παράθυρο ευκαιρίας το οποίο μπορεί να μην επαναληφθεί και οι ηγέτες των Σκοπίων ξέρουν ότι αν χάσουν αυτή την ευκαιρία δεν θα μπορέσουν εύκολα να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Αυτό είναι και το κλειδί στην πόρτα της ε, ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα για τον διάλογο τώρα <clears throat> μεταξύ Βελιγραδίου και Πριστίνες. Είναι απαραίτητο να έχουμε μια νυφάλια προσέγγιση, να αντιμετωπίσουμε τεχνικά προβλήματα. Όλα είναι πολιτικά, αλλά τα τεχνικά προβλήματα τα οποία φύγουν την καθημερινότητα των πολιτών πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι στιγμή για τα μητρώα κτλ. Όλα αυτά είναι μικρά βήματα. Θα πρέπει να έχουμε μια λογική φιλοδοξία να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε όσο μπορούμε <clears throat> όσο είναι διατεθειμένοι να επιτύχουν οι εταίροι από το Βελιγράδι και την Πριστίνα. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια θετική ατμόσφαιρα ώστε να πιστεύουν και οι δύο πλευρές ότι υπάρχει ένας αρρηκτός διάβλος επικοινωνίας που θα είναι χρήσιμος και να συνεχίσουν να συμμετέχουν σε αυτό το διάλογο. Αυτό είναι ο στόχος μας και αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Η κυρία Πακ <clears throat> για τη Βοσνία Ζεχοβίνη. Δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι και εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος από την κατάσταση αυτή με τα, με τα αποτελέσματα αυτής της ε, διαδικασίας. Δεν μπορεί κανείς να αποκλείει από την <clears throat> κυβέρνηση πολιτικά κόμματα τα οποία στην εθνοτική τους κοινότητα εκπροσωπούν την πλειοψηφία των ψηφοφόρων. Χρειάζεται να υπάρχει σε όλα τα επίπεδα ισχυρή κυβέρνηση στη Βοσνία Ζεγοβίνη, αν θέλουμε μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρο να εφαρμόσει τι απαραίτητε μεταρρυθμίσει και να τι περάσει και από το Κοινοβούλιο τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Η ισχυρή παρουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι θα έχουμε ένα εκπρόσωπο, τον επικεφαλή τη αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίο θα είναι και ο νέο ειδικό εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί. Θα στείλουμε λοιπόν προσωπικό και θα δώσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση για να υπάρχει αυτή η παρουσία και ο υψηλός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αντιμετωπίζει τα πολιτικά θέματα χωριστά από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, χρειαζόμαστε περισσότερο, περισσότερη χρηματοδότηση, χρηματοδότηση είπε, από το πρόγραμμα ΕΙΠΑ της τάξης των 100 εκατομμυρίων το χρόνο και να έχουμε διαδικασίες όπως η απαγόρευση προξενικής θεώρησης ή το πάγωμα των στοιχείων ενεργητικού αυτών οι οποίοι δεν συμμορφώνονται. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια νέα συμφωνία Dayton Sin. Θέλουμε οι Βόσνοι να μιλούν με ενιαία φωνή, αλλά δεν το κάνει καν και η διεθνής κοινότητα εναντί τους. Τα συμπεράσματα των Υπουργών Εξωτερικών το Μάρτιο ήταν ένα σαφέ μήνυμα για το ποια είναι η στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα, την περιμένουν από τη Βοσνία Ζεγοβίνη και επομένω θα πρέπει και αυτοί να γνωρίζουν τι περιμένουν από εμά. Είναι μια πρόσκληση για συζήτηση και με άλλου διεθνεί εταίρου. Ο στόχο μα θα πρέπει να είναι η σαφήνεια. Αυτό το οποίο θέλουμε λοιπόν να επιτύχουμε είναι αυτή η σαφήνεια. Στο κοσυφοπαίδιο. ε, ανασυγκροτούμε πάλι την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να υπάρχει μεγαλύτερη ορατότητα στην παρουσία μας και καλύτερη ποιότητα στο ρόλο μας. Συνεχίζονται οι συζητήσεις ακόμα μεταξύ των 100 μελών για το πώς θα το πετύχουμε. Αναφέρθηκε η παρατήρηση των εκλογών. Εγώ υποστηρίζω <clears throat> την παρακολούθηση των εκλογών γιατί μας δίνει πληροφορίες σε πρώτο χέρι. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε στα χέρια μας τις ευθύνες της πολιτικής τάξης για αμερόληπτες και καθαρές εκλογές. Αυτό είναι δική τους ε, αρμοδιότητα και όχι δική μας. Πάλι για τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Εμείς προχωρούμε στα παρασκήνια πολλές φορές με ήρεμο τρόπο και όχι με ε, την πανοκρουσίες να βελτιώσουμε τα πράγματα ώστε να μπορέσει η κυβέρνηση εκεί να δώσει απάντηση στις προσδοκίες μας. Χρειαζόμαστε πραγματικά μια ισχυρή κυβέρνηση για την Πουδουγουμού. Το θέμα του ονόματος είναι το κύριο θέμα το οποίο πρέπει να επιληθεί, αλλιώς δεν θα μπορέσει να υπάρξει καμία πρόοδος. Και εμεί θέλουμε φυσικά να υπάρξει πρόοδος. Για τον πρόεδρο του Κοσφοπεδίου δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο από ό,τι ξέρετε. Αυτό, είναι το... Αυτό που είναι απαραίτητο είναι να βρεθεί μια συνταγματική Λύση και να σταματήσει η συνταγματική αυτή η κρίση. Να υπάρξει μια διαδικασία που θα γίνει μέσα από τους ίδιους του θεσμούς του και συμμετοχή των Σέρβων στην πολιτική ζωή του κωσφοπεδίου. Είναι και αυτό το τμήμα του διαλόγου και τμήμα της προσπάθειάς μας να αναπτύξουμε διάλογο με το Βελιγράδι γιατί και το Βελιγράδι είναι τμήμα της διαδικασίας, είναι μέσα σε μια διαδικασία ένταξης και όλες οι δραστηριότητές τους, όχι μόνο η τεχνική εφαρμογή του κεκτημένου, αλλά η γενική στάση του ε, Βελιγραδίου σε σχέση και με τους γείτονές, γείτονές του παίζει ρόλο στην εκτίμησή μας. Κυρία Λούνατσεκ, εγώ χαίρομαι για τη συνάντηση αυτή με τους Σέρβους δήμαρχους από το Κοσμοπέδιο και τη δυνατότητα επικοινωνίας όχι μόνο σε κεντρικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο για την ε, απογραφή. Είμαστε σε επαφή με τους συνομιλητές μας ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα διενεργηθεί αυτή η απογραφή και θα τηρήσει τα αναμενόμενα από εμά. Θα πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος στο κοσχοπέδιο, δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Ίσα ίσα μπορούν να δείξουμε τον τρόπο αυτό το επικοδομητικό τους πνεύμα και να δείξουν τη θέλησή τους για να συνεχίσουν αυτήν την ε, διαδικασία είναι και η λυδία λίθος για να μπορέσουμε και εμείς να δούμε ότι υπάρχει ένα επικοδομητικό πνεύμα. Από τη στιγμή που υπάρχει πρόοδος επικοδομητική στο διάλογο αυτό θα βελτιώσει ιδιαίτερα και το κλίμα και το κύρος του κοσμοπεδίου σε σχέση με τους διεθνείς εταίρους τους. Η επιτυχία λοιπόν στη διαπραγματεύση είναι πάντα θετική. Για την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμείς ε, βρίσκουμε τώρα μια προσωρινή λύση που θα καλύψει το διάλογο το διάστημα μέχρι, την, μέχρι τον διορισμό του επόμενου αντιπροσώπου. Ο στόχος μας είναι ότι θα έχουμε πάντα μια συνεχή παρουσία επιτοπίως για να συνεχίσουμε το έργο μας. Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για χρονικό ορίζοντα, γιατί συνεχίζονται οι συζητήσεις μεταξύ των κρατών μελών και δεν ξέρουμε και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας συζητήσεων. Νομίζω ότι μέσα σε δύο ή τρει μήνε θα έχουμε μια σαφήνεια σε σχέση με τι μελλοντικέ δομέ εκεί. <clears throat> Κροατία και η κοινή γνώμη. Ήμουνα μαζί με τον πρόεδρο Μπαρόσο στην επίσκεψή του και αυτό που είδα εκεί είναι μια σαφής προσήλωση από όλου του κυβερνητικού θεσμού και από τα πολιτικά κόμματα για να εργαστούν, να εκπληρώσουν τα υπόλοιπα κριτήρια ώστε να μπορέσει να ενταχθεί η Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το γενικό κλίμα είναι επικοδομητικό εκεί. Αναγνωρίζουν όλοι ότι δεν είναι εύκολο να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά εγώ εντυπωσιαστικά από τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η πολιτική ηγεσία. Κύριε Τάνοκ, το Μαυροβούνιο. Δεν θέλω να μιλήσω εδώ για χρονοδιάγραμμα έναρξης διαπραγματεύσεων. Για το Μαυροβούνιο όμως είμαστε σε καλή κατάσταση, γιατί το Μαυροβούνιο έχει κάνει ακριβώς αυτό το οποίο περιμένανε περιμέναμε από αυτού, ξέρουν ποιε είναι οι κύριες προτεραιότητε, τι έπρεπε να επιτύχουν και υπάρχουν συνεχεί εκθέσει πρόοδου κάθε μήνα για την πρόοδο που επετελέστη. Και η επόμενη έκθεση πρόοδου τη Κομισιόν τον Οκτώβριο θα μα δώσει μια σωστή εικόνα τη κατάσταση. Αλλά η δική μου εντύπωση από την επίσκεψή μου εκεί ήταν πολύ θετική γιατί η νέα κυβέρνηση είναι πράγματι δεσμευμένη και προσιλωμένη στη διαδικασία αυτή ένταξη. Για την Πουδουγού μου απήντησα ήδη και για το κοσυφοπαίδιο η διχοτόμησή του δεν είναι μια λύση η οποία υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την έκθεση Μάρτη τώρα για το εμπόριο οργάνων. Έχουν ξεκινήσει οι έρευνες, έχουμε έρθει σε επαφή με τον κύριο Μάρτη από το Συμβούλιο της Ευρώπης πολλές φορές. Ήμουν σε επαφή με τον επικεφαλής της Γιούλεξ, δεν υπάρχει πρόβλημα στελέχωσης με ανθρώπινο δυναμικό και με οικονομικούς πόρους. Υπάρχει μια ειδική μονάδα η οποία θα αντιμετωπίσει αυτές τις ε, έρευνες και εργαζόμαστε επίσης και για την προστασία των μαρτύριων. Είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να ξέρουμε πόσο σημαντική προστασία θα χρειάζεται, πόσοι μάρτυρες θα καταθέσουμε. Αλλά θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανάγκες όταν παρουσιαστούν. Και γενικότερα για το θέμα της ε, κόπωσης, διεύρυνσης, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο στα Δυτικά Βαλκάνια. Και δεν νομίζω ότι μόνο το Μοντενέγκρο είναι πετυχημένη χώρα από τα Δυτικά Βαλκάνια. Κάθε άλλο. Αν δεν ήταν η διαδικασία <clears throat> ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατάσταση θα ήταν πολύ πιο ζωφερή. Οι χώρες αυτές ξέρουν ότι έχουν αυτή την προοπτική, ξέρουν ακριβώς τι περιμένουμε από αυτές για να είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν καιρό. Αυτό το οποίο πρέπει να πράξουμε είναι να είμαστε πάρα πολύ σαφείς για τους όρους που θέτουμε και να κρατήσουμε πάντα σε επίπεδο του εφικτού το στόχο αυτό της ενσωμάτωσης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάλι για τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Όπως είπα προηγουμένως, πρέπει να υπάρχει σαφήνεια για το ρόλο της διεθνή κοινότητα και για την παρουσία που θα έχουμε εκεί. Και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών του Μαρτίου πηγαίνουν προ τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα θα πρέπει να συμφωνήσουμε για τις προποθέσει να καταργηθούν σταδιακά οι αρμοδιότητες του υπάτου εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποδοθούν στο πολιτικό σύστημα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Αν δεν λειτουργεί σωστά το σύστημα αυτό, σημαίνει ότι η διεθνή κοινότητα δεν έχει δράσει σωστά στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Δεν πρέπει λοιπόν να ρίξουμε σε αυτού μόνο το φταίξιμο, θα πρέπει να κατανοήσουμε τι έχουμε κάνει και από τη δική μα πλευρά. Είπα για τι εκλογέ του Πρόεδρου του Κωσυφοπεδίου, Αλβανία, και αυτό το απήντησα περιμένουν όλοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση καλές προοπτικές και σαφήνεια. Δεν πρέπει να μετακινήσουμε τα τέρματα του ποδοσφαιρικού γηπέδου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Πρέπει ο στόχος να είναι απτός και επιτεύξιμος όπως στην περίπτωση της φιλελευθεροποίησης των προξενικών θεωρήσεων. Εκεί ήταν σαφές το, το δικό διάγραμμα. Και τώρα η Κροατία και το Μαυροβούνιο ξέρουν ακριβώς πού βρίσκονται και ποιε είναι οι απαιτήσει για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Και έτσι κρατιούνται στο σωστό δρόμο. Νομίζω ότι απήντησα και το ερώτημα για τις προοπτικές. Οι διεθνείς εταίροι στη Βοσνία Ζεγοβίνη, ιδίω οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία έχουν δείξει την εκτίμησή τους για τα συμπεράσματα του Μαρτίου, γιατί πολλές φορές είχα ρωτηθεί ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποια είναι τα εργαλεία που έχετε στη διάθεσή σα ποια είναι τα και στις στρατηγικές σας στον τομέα αυτό, με τα συμπεράσματα θα έχουμε δώσει μια απάντηση. Και <clears throat> μπορούμε επομένως να συζητήσουμε με τους διεθνείς εταίρους μας για το μέλλον αυτής της Διεθνούς Επιτροπής στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Θα χρειαστεί χρόνο γιατί αυτοί οι εταίροι και οι ρωσικοί... Ομοσπονδία επίση έχουν τι δικέ του προσδοκίε για το τι πρέπει να γίνει στη Βοσνία Ζεγοβίνη, αλλά νομίζω πρέπει να κρατήσει ηγετικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση και με, ε, με τα συμπέρασμα του Ματίου δείξαμε ότι αυτή είναι και η δική μα φιλοδοξία. Και πιστεύω ότι έχω απαντήσει όλα τα ερωτήματά σα Για τον κύριο Μποστινάρου, στι συζητήσεις με του εταίρους μα από την περιοχή είναι σημαντικό να δίνουμε ευρωπαϊκά μηνύματα, να τους ευρωπαϊκοποιήσουμε και όχι να χρησιμοποιούμε τις εσωτερικές τους διαμάχες. Πρέπει τα μηνύματα λοιπόν τα οποία έρχονται από τις Βρυξέλλες να είναι σαφή και να μην, τους να περιμένουμε ότι... να περιμένουμε ότι αυτοί θα λειτουργούν σαν και εμάς και όχι με διαφορετικό τρόπο. Ευχαριστώ. Οι συνάδελφοι εκτίμησαν την ακρίβειά σας και την πληρότητα των απαντήσεών σας. Δεδομένων των χρονικών περιορισμών μας, τα πήγατε πραγματικά εξεχόντως καλά. Ευχαριστούμε για το έργο που φέρατε σε πέρας και τα περιμένουμε κάποιες εβδομάδες ή και μήνες για τις τελευταίες εξελίξεις που θα μας δώσουν την ευκαιρία να εκφράσουμε και την ευαισθησία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τώρα θα περάσουμε στην ψηφοφορία, η οποία θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά. Chairman, can we uh, start? Πρόεδρε, μπορούμε να ξεκινήσουμε, γιατί έχω να παραστώ και σε άλλες συνεδριάσεις. My answer to the question... Η απάντησή μου στην ερώτησή σας είναι μάλιστα κύριε, αμέσως. Ας προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Θέλω να βάλετε όλοι τις κάρτες σας στη σχισμή και θα ξεκινήσουμε με την έκθεση του κυρίου Αλμπερτίνη. Είσαστε όλοι έτοιμοι. Τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36. Ποιοι είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Θα πρέπει να ελέγξουμε. Η 36. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 37. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην 50. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 51. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 52. Ναι, μπορούμε να ελέγξουμε, αν θέλει. Για την 51. Πέρα της, της ψηφοφορίας. 41 προς 18. Απορρίπτεται. Η 52. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 53. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Θα πρέπει να ελέγξουμε. Επομένως... Η 54. Η 54 ψηφίζουμε για την 54. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 55. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 6. Ποιοι είναι υπέρ. Α. 6. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα περνούμε στην 59. Ποιοι είναι υπέρ? Συγγνώμη. Τι συμβαίνει με την, με την 56, τι έγινε με την τροπολογία 56. Ερώτηση του κυρίου Νταφ. Ε, εγκρίθηκε η 53. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, λέει ο κύριο Νταφ. Ε, εντάξει, 59. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 60 υπέρ, κατά. Αποχές, θα πρέπει να ελέγξουμε για την 60. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 35 κατά, 30 υπέρ. 61. Ποιοι είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60... Η 63. Ποιοι είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 67 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 68 υπέρ, Κατά. Εγκρίνεται. 69 υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνούμε στην τροπολογία 81. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, θα πρέπει να ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 81. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 82 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 84 υπέρ, κατά, θα πρέπει να ελέγξουμε. Για την 84 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 32 ε, κατά, 31 υπέρ. Περνούμε λοιπόν στην τροπολογία 85 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 86 υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 89. Αυτή ήταν η 88. Α, ελέγχουμε για την 88. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 32 κατά 26 υπέρ. 89. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συγγνώμη. Αποχές δεν είπα. Εντάξει. Θα Εντάξει να ελέγξουμε. Ελέγχουμε για την 89. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Α, 31-31. Δεν το περίμενα αυτό. Άρα απορρίπτεται. Παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου. Εκτός μικροφώνου. Έκανα λάθος όταν ψήφισα. Ε, ήδη, ήδη είχε απορριφθεί, οπότε δεν ήταν ανάγκη να μας το πεις. Ευχαριστώ πολύ. 90. Υπέρ της 90. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Επομένως, περνούμε στην 103. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 101. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 104. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 105. Υπέρ, κατά, Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά θα ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 105. Mm. Απορρίπτεται με δύο ψήφους, 33 ε, έναντι 31. 106 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά. Το ίδιο. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 115. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Εκατόν υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 13 σε 3 μέρη. Το πρώτο μέρος υπέρ. Με συγχωρείτε. Αντιτίθεμαι στην ψηφοφορία της προφορικής τροπολογίας που, υπέβαλαν η ΕΛΚ, που υπέβαλε το ΕΛΚ. Αν επιμένουν θα πρέπει να μας φέρουν την τροπολογία για να μπορέσουμε να την συζητήσουμε σωστά. Επομένως, ε, θα πρέπει να μας εξηγήσουν την προφορική τροπολογία. Εκτός μικροφώνου. Όχι, όταν υπάρχει αντίθεση, ένσταση, ακόμα και από ένα μόνο βουλευτή, δεν πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία η τροπολογία. Εντάξει. Ψηφίζουμε τώρα την συμβιβαστική τροπολογία 13, το πρώτο μέρος. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το τρίτο τμήμα υπέρ Όχι, για το τρίτο μέρος, επειδή το δεύτερο μέρος δεν θα τέθει σε ψηφοφορία λόγω της ένστασης. Τρίτο μέρος λοιπόν, υπέρ, κατά, νομίζω ότι έχει απορριφθεί. Εντάξει, αν θέλετε να ελέγξουμε, θα το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρα της ψηφοφορίας. Α, πόσο δίκιο είχατε. Όπως πάντα. Εντάξει. Περνούμε τώρα στην 138. Ε, 138 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 139 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Επομένως, περνούμε στην 148 υπέρ, κατά, Πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 148. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 151 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 152 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 153 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. έλεγχος για την 153. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται λοιπόν. 154 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα ελέγξουμε. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 154. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και έτσι περνούμε στην 169. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 170 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 171 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 172 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 173 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 174 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 175 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 176 υπέρ, Θα ελέγξουμε. Έλεγχος για την 176. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Έχουμε μία παραπάνω ψήφο, αλλά εγκρίνεται. 177. Υπέρα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 180 υπέρ, κατά, άποχες εγκρίνεται. 178 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 179 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 183 υπέρ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 192 υπέρ. Κατά. Θα πρέπει να ελέγξουμε παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 192. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 193 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 186 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 186. Πέρας της ψηφοφορίας. και ο νικητής είναι εγκρίνεται. 187 υπέρ. Κατά. Πάλι πρέπει να ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 187. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 188 υπέρ. Κατά. Ναι, η ίδια πλειοψηφία. Εγκρίνεται. 189 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Εκα... Ε, καταπίπτει 190. Εάν υιοθετηθεί... Εάν εγκριθεί 186, αγκρίθηκε 186. Συμβιβαστική τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 18. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 200. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 204. Υπέρ, κατά, το ίδιο, εγκρίνεται. 206. Υπέρ, Απορρίπτεται. 207. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 209. Ε, Υπέρ. Συγγνώμη, 208 λέει ο μιλητής. 208. Υπέρ. Κατά. Θα το ελέγξουμε για την 208. Ε, Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίφθηκε. 209 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 210 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 211 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε 2.18. 218 υπέρ, κατά, αποχές, πρέπει να ελέγξουμε. Για, την 218 αρχίζει η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται λοιπόν. 219 υπέρ, κατά, Αποχές. Νομίζω ότι είναι η ίδια πλειοψηφία, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 219. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2 Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 228. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 229. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 233 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 234 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 235 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 236 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 237 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 238 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 22 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Επομένως, περνούμε στην... Ναι, στην 244 υπέρ, κατά, Αποχές νομίζω πρέπει να το ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία για τη 244. Δουλεύει, λειτουργεί, εντάξει, εγκρίνεται. Περνούμε στην συμβιβαστική τροπολογία 23, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 250 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οπότε, περνούμε στην 259 υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. 260 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 261 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 262 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 263 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 264 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 265 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 266 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 267 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 268 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 268. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ο κύριος, κύριε Βαν Βόρντεν, ψηφίσατε και την ίδια την τροπολογία σας. Εντάξει, Πέρασε τη ψηφοφορίας. Ναι, ψηφίσατε, εντάξει. Εγκρίθηκε. 269 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 270 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 271 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 272 υπέρ, κατά, θα πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη 272. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 273 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στη 10. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. εντάξει, πάρει. Who is against? Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ, όχι 17, 18. 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19 υπέρ, Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας ελέγξουμε καλύτερα. Για τη 19. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αριθμός 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Εντάξει, για την αριθμός 4. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τώρα, γνωμοδοτήσει τη Επιτροπή Προπολογισμών. Γνωμοδότηση, μάλλον τη Επιτροπή Προπολογισμών. Οι σχετικέ τροπολογίε 1 συν 3 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνονται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 6 και 7 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οι άλλες παράγραφοι τώρα. 4, 5, 8 και 10 είναι κατά ο εισηγητής. Οπότε τις ψηφίζουμε μαζί. 4, 5, 8 και 10. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα για την τροποποιημένη έκθεση. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορίας. Κύριε Αλμπερτίνη, μεγάλη επιτυχία. Ο κύριος Μέρ το λόγο. Παρακαλώ. Ο κύριος Μαγιώρα, ευχαριστώ. Εμείς θα υποβάλουμε έκθεση μειοψηφίας, η ομάδα μας. Καλώς, λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε. So here uh, Καλώς. Εδώ θα χρειαστεί, ναι. Να επιβραδύνουμε. Γιατί χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις στην προφορική αριθμός 5 για παράδειγμα τροπολογία, διότι εκεί υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις που θέλει να μας κάνει ο εισηγητής. Αλλά κύριε Κόπα θέλει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να αποσύρω τις τροπολογίες μου 9, 32, 55 και 2009. 209. Oh. Α, τι είπα λάθος, λάθος το είπα λέει η κυρία Κόπα. 9 ήθελα να πω. Ε... So it's 9. 9, 32, 55 και 209, λέει ο πρόεδρος. Εντάξει. Να το σημειώσουμε. 9, 32, 55 και 2009 είπατε. Εντάξει. Καλώς. Είμαστε έτοιμοι. Τροπολογία αριθμό 6. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. απόχέ, Απορρίπτεται. 7. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Συμβαστική αριθμό 1. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική αριθμός 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία αριθμός 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά Α, είναι δικιά μου. Εντάξει, λέει ο πρόεδρος. Εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά θα ελέγξουμε. Για την 34 παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 35 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ, κατά, Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά σε λέξουμε καλύτερα. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 39. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. Τρεις παραπάνω από τους σοσιαλιστές. Εγκρίνεται με πέντε ψήφους διαφορά. Οι τρεις όμως είναι παραπάνω, ε? οπότε βρείτε τα μεταξύ σας ποιοι ψηφίζουν και ποιοι όχι. Πέντε είναι η διαφορά, οπότε και να βγάλουμε τις τρεις, πάλι το ίδιο αποτέλεσμα έχουμε. Πάντως τρεις ψήφοι από τους σοσιαλιστές πρέπει να φύγουν. Βρείτε τα. Λοιπόν, ψηφίσαμε την 39 μόλις τώρα. Και τώρα περνάμε στην 40. 34. Θα ελέγξουμε για την 34 αφού θέλετε. Εντάξει, για την 34. 34. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρες ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εντάξει τώρα. Είναι εντάξει τώρα και η ψηφοφορία και όλα. Κάποιοι αλλάξανε γνώμη προς το καλύτερο, λέει ο πρόεδρος. Συνεχίζουμε και ψηφίσουμε τώρα τη 40. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική αριθμός 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 και 50 που είναι ίδιες. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Απορρίπτονται. Είναι ξεκάθαρο, αλλά αν πραγματικά θέλετε, θέλετε. Ωραία. Να ελέγξουμε για την 49 και 50. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορία. Ε, σας είπα, δεν είχε νόημα. 51. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 54. Σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Να για το δεύτερο τμήμα παρακαλώ. Ψηφίστε για το δεύτερο τμήμα της 54. Πέρας της Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τέταρτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε για το τέταρτο τμήμα της 54. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Και εδώ δεν έχουμε παραπάνω ψήφους από κανέναν. Άρα αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Παρέμβαση εκτός μικροφώνου ζητάτε πάρα πολλά, απαντάει ο Πρόεδρος. 56 τώρα. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά να ελέγξουμε καλύτερα την 56. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία των αριθμών 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στην 62. Όχι. Α, όχι. Πρώτα 58 και 59. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61, όχι. 62 τώρα. Ε, όχι το 61, α, 61, 61, υπέρ της 61. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 62. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται νομίζω, αλλά να ελέγξουμε. 62, ελέγχουμε, ψηφίστε. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία αριθμός 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 70 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προσθήκη από ό,τι μου λένε είναι. Για προσθήκη στην προφορική τροπολογία αριθμός 72. 71 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 73 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 75 υπέρ, κατά, εγκρίνεται νομίζω, αλλά να ελέγξουμε καλύτερα για την 75. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Ναι, εγκρίνεται. 76 και 100 έχουν ε, αποσυρθεί. 77 τώρα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 4 τώρα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην 91. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Την ψηφίσαμε την προφορική 4. Απαντάει ο πρόεδρος, ε, παρέμβαση εκτός μικροφώνου. 91 τώρα υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 99 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 101 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να ελέγξουμε καλύτερα για την 108. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη φοφορίας. Εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 110 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 112 υπέρ, κατά, απορρίπτεται νομίζω, αλλά σε ελέγξουμε καλύτερα. Την 112 παρακαλώ, ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 113 τώρα σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ. Κατά. Να έλεγξουν. Ξεκινάει η ψηφοφορία. 113 πρώτο τμήμα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με μία ψηφοδιαφορά χωρίς παραπάνω ψήφους. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Α, να ελέγξουμε. Καλά. Δεύτερο τμήμα, ελέγχουμε. Ψηφίστε. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Το ξέρατε, το ξέρατε. Θα μπορούσατε να μου το είχατε ψιθυρίσει για να μου το φωνάξετε έτσι. Να μου το πείτε διακριτικά. 114 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε για την 115 ηλεκτρονικά. Άλλη μία ψήφος χρειάζεται. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Απορρίπτεται. Και πάμε στη συμβιβαστική αριθμός 5. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 122. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 128, όχι. Συμβιβαστική 7 τώρα, υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 136 τώρα, υπέρ. Κατά. Αυτό είναι κομματική πειθαρχία, λέει ο πρόεδρος. Αποχές απορρίπτεται. 137 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι γκρίνεται 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 140 υπέρ κατά Απορρίπτεται. Ναι. Δεν θα ελέγξουμε. Απορρίπτεται. 141. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Για την 142 θέλετε το λόγο κύριε Λτιέρη. Α, μετά την 142. Ωραία, 142 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τώρα ο κύριος Χολτιέρη θέλει κάτι να πει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να προτείνω μια προφορική τροποποίηση στην παράγραφο 30 που λαμβάνει υπόψη την τροπολογία 209 που αποσύρθηκε και πρόκειται για μια μικρή αλλαγή όσον αφορά την αλληλεγγύη και τις πολιτικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις θέλω να πούμε ότι υπενθυμίζει ότι η αμοιβαία αρρωγή είναι η υποχρέωση για την αλληλεγγύη σε περίπτωση που υπάρξει εξωτερική επίθεση σε οποιοδήποτε χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να μην αντιβαίνει στην ρύθμιση του ΝΑΤΟ για το σεβασμό και την δετερότητο ορισμένων ε, χωρών μελών. Ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή αυτή η δετερότητα. Παρέμβαση εκτός μικροφώνου. Δεν ακούμε. Ποιο είναι κατά τη τροποφορικής αυτή τη τροπολογίας. Εγώ αντιστήθαμε στην τροποφορική τροπολογία. Εντάξει, ταξιαρχέ μου. Τότε δεν ισχύει νομίζω ότι δεν μπορούμε εμεί τώρα να αλλάξουμε τη στρατηγική, την αρχιτεκτονική στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πολύ παράδοξο. Είναι πιο μεγάλο, λέει ο κύριο Φανόρντεν. 133 υπέρ, κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. 1,44 υπέρ, κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. 1,45 υπέρ, κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. 146 υπέρ, κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά σε ελέγξουμε 146 ηλεκτρονικά <clears throat> άρχεται πέρας εγκρίνεται με μία μόνο ψήφο πλειοψηφία 147 υπέρ κατά αποχές δεκτή 148 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 149 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 154 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 153. Όχι, εκπίπτει. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 158. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 100... Προφορική τροπολογία 5 τώρα. Υπέρ. Κατά. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Η 158 δεν εγκρίθηκε. 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. θέλετε να εξηγήσετε στο κοινό περί τίνος πρόκειται. Τεχνικό είναι το πρόβλημα, λέει ο κ. Γκουαλτιέρη, με την προφορική τροποποίηση 5, οι τροπολογίες 163, 164, 165 και 167 εκπίπτουν. Μόνο την 162 πρέπει να το ψηφίσουμε γιατί είναι τυπική αλλαγή και μετά να πάμε στην 166. Στην προφορική 6 μάλλον. Η 162 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Προφορική υπαριθμών 6 του εισηγητή. Ψήφι υπέρ. <clears throat> Κατά. ποχές Δεκτή. 168 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 169 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 170 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 171 υπέρ

κατά αποχές δεκτή. 1,77 υπέρ. Να ελέγξουμε πρώτα την 176. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία επαλήθευσης. Πέρας. Απερίφθη σαφώς. 177 υπέρ. κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 9 Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 181. Υπέρ. Κατά. Αποχές πρέπει να ελέγξουμε. Έλεγχος ηλεκτρονικός για την 181. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απέριπτε. 182 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 183 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 184 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 185 υπέρ κατά. Ας ελέγξουμε την 185 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 187 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 188 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 189 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 190 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 193 υπέρ κατά αποχές δεκτή 194 υπέρ κατά αποχές δεκτή 195 υπέρ κατά Αποχές δεκτή 196 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Να ελέγξουμε για την 196. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Κάποιοι δεν καταλάβανε και δεν... Ναι, ναι. 197 υπέρ κατά δεκτή 198 υπέρ κατά αποχές δεκτή 199 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 200 με 202 που είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 203 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 204 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 205 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά <clears throat> αποχές απορρίπτεται 207 υπέρ κατά αποχές δεκτή 208 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 210 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 211 υπέρ κατά από... πρέπει να λέξουμε. άρχεται η ψηφοφορία για την 211 πέρας απορρίφθηκε 212 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 213 υπέρ <clears throat> κατά αποχές απορρίπτεται. 214 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 215 όχι. 216 μάλλον υπέρ κατά αποχές έλεγχος για 216. Άρχεται η ψηφοφορία. Καλησπέρας. Εγκρίνεται. 2.17 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2.18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.19 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. 220. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. <clears throat> Απορρίφθηκε. 2.21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. τεκτή. 2-2-4 <clears throat> υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2-2-5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2-2-6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2-2-7 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της 227 άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 2.28 όχι δεν ψηφίζουμε, γιατί εγκρίθηκε το δεύτερο τμήμα. 2.29 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. 2.30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.31 εκπίπτει, όχι δεν εκπίπτει, ψηφίζουμε 2.31 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θα ελέγξουμε τη 2.35 Πέρας. Εγκρίθηκε. 2.36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 ναι ναι φαινόταν από το πρωί 2.37 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 2.39 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 2.38 υπέρ. Όχι, όχι, εγκρίθηκε η προηγούμενη. 2.40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.41 υπέρ. Κατά. Αποχές. <clears throat> εγκρίνεται. 2.43 υπέρ. Κατά. Σχές. Ας ελέγξουμε. 2.43 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. 2.44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.45 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Προφορική 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 2.46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.47 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.49 υπέρ κατά Σηκώστε τα χέρια σας. Έλεγχος στη 249. <laughs> Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.50 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.51 υπέρ. Κατά. <clears throat> Αποχές απορρίπτεται. 2.52 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2.53 σε δύο τμήματα, τμήμα 1 υπέρ κατά. Θα ελέγξουμε πρώτο τμήμα της 253. Πέρας. <coughs> Εγκρίθηκε με δύο ψήφους διαφορά. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Το ίδιο αποτέλεσμα νομίζω. Εγκρίνεται. 2.54 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.55 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για τη 255, μάλιστα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. απέριπτε <clears throat> με τρεις ψήφους διαφορά. Λοιπόν, 2.56 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 2.57 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 2.58 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική 8 του εισηγητού ψήφι υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.59 υπέρ, κατά απορρίπτεται 2.60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και αυτή 2.61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.63 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 2.64 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.65 υπέρ 265 λέμε. Υπέρ. Κατά. Α, ελέγχουμε γιατί 265. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Με μία ίσχυνη ψήφο εγκρίνεται. 266 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 267 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 2,60 τελευταία σελίδα 2,68 <clears throat> υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2,69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2,70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2,71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αλλά θα ελέγξουμε ούτως ή άλλω 2-71. Άρχεται η αλλω 271 αρχεται ελέγχου. ελεγχου περα τη αυτή τη ψηφοφορία ελέγχου. Απορρίπτεται. 2.72 υπέρ. Κατά. αποχε Απορρίπτεται. 2.73 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 2.74 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε 2.74 έλεγχος πέρας τις ψηφοφορίες. απορριφθήκε 2.75 υπέρ κατά αποχές δεκτή 276 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. 276. Αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Ισοψηφία απορρίπτεται, δύο όμως βουλευτές δεν ψήφισαν, κράτησαν στάση αποχής. Αυτοί εκεί πέρα τους βλέπω στο βάθος. Η κυρία Λέζον και ο κύριος Μάιερ. Απορρίπτεται την πάση περιπτώσει. 2,77 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2,78 υπέρ. Κατά. Αποχές δεχτεί. 2,79 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 2.80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.81 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.82 <clears throat> υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.83 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.84 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ένα. υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δύο. υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τρία. υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τέσσερα, πέντε μάλλον. Τέσσερα. υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τελική ψηφοφορία. Παρακαλώ. Πέραση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Συγχαρητήρια κύριε Γουαλτιέρη. Κυρία Λέζινγκ, έχετε το λόγο. Και σε αυτή την έκθεση η πολιτική μου ομάδα θα καταθέσει μια minority report, μια μειοψηφική έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. τελευταία ψηφοφορία. Τελευταία ψηφοφορία. Όσοι θέλουν να φύγουν, να μην φύγουν. Τροπολογία υπαριθμών Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 6 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Σε δύο τμήματα. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 11. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική υπαριθμών 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ εκπίπτει 22 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά θα ελέγξουμε για την 22 Πέρας προφορίας. Εγκρίνεται. Πριν από την τελική ψηφοφορία, ο κ. Προτάσιβιτς θέλει να κάνει μια πρόταση. Έχετε τον λόγο κύριε Προτάσιβιτς. Ευχαριστώ. Θέλω να πω στα μέλη του ΕΛΚ, τώρα μπορούμε να ψηφίσουμε υπέρ. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίστε λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ένας αγνοούμενος. Λείπει μάλλον μία ψήφος. Πέρασε ψηφοφορίες. Εγκρίνεται και συγχαρητήρια στην κυρία Λέζιν. Κύριε Αλμπερτίνη, σας ξαναδίνω τη θέση του Πρόεδρου. It's not in my hands any longer. It's in Mr. Albertini's hands. Δεν είναι πια στα δικά μου χέρια. Ε, τώρα εναπόκειται στον κύριο Αλμπερτίνη.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 Ε, <clears throat> eh, Συνάδελφοι, να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το 15, που αναφέρεται στην πρώτη ανάγνωση της έκθεσης του Jeffrey Van Orden. Η έκθεση αφορά τις ε, προκλήσεις ε, και ό,τι ισχύει στον έλεγχο των ναρκών. Θα δώσω κάποια, να σας ενημερώσω για δύο-τρία πράγματα πριν δώσω το λόγο στον κύριο Βαν Όρντεν. 3 Μαΐου είναι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών και η συζήτηση επί των τροπολογιών θα γίνει στις 9 Μαΐου. Η ψήφιση προβλέπεται για τις 24 Μαΐου. Έχετε το λόγο κύριε Φανόρτεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω ότι γενικά δεν θα δημιουργηθούν και πολλές διαφωνίες σε σχέση με αυτήν την έκθεση. Νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ των συναδέλφων σε όλο το κοινοβούλιο. Δεν είναι μια μονόπλευρη έκθεση. Έχουν περάσει 12 χρόνια από τότε που η Σύμβαση για τις Νάρκες τέθηκε σε ισχύ. Θα θυμάστε η σύμβαση υπογράφτηκε για να απαγορεύσει την παραγωγή και χρήση και κατοχή ε, χερσαίων ε, ναρκών. 166 χώρες έχουν υπογράψει τη σύμβαση μέχρι στιγμής. Ε, πέρα από διάφορες ανησυχίες, θεωρήσαμε ότι είναι καλό να ξαναδούμε το θέμα της απενεργοποίησης των ναρκών και να δούμε ποιοι είναι οι φορείς που συμμετέχουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει πάρα πολύ, τα κράτη-μέλη, ο Καναδάς και οι Ηνωμένε Πολιτείε ιδίω. Πολλοί από εμά συμβάλαμε στην σχετική διακήρυξη και συμμετείχαμε στην χρηματοδότηση των ε, ενεργειών αποναρκοθέτησης αλλά εξακολουθούμε, εξακολουθούν να σημειώνονται θάνατοι από τις νάρκες αυτές και να χορηγούνται πόροι ε, για την αφαίρεσή τους. Ε, η έμφαση είναι στις νάρκες κατά προσωπικού όλος ιδιαίτερος σε αυτήν την κατηγορία. Επίσης στα εκρηκτικά υπολείμματα ναρκών και περιλαμβάνει όλα τα πυρομαχικά καθώς και τις βόμβες διασποράς, τις νάρκες διασποράς. προσπαθούμε να βοηθήσουμε, υπάρχουν ε, σωστά κίνητρα και δεν χρειάζεται να αυτομαστιγωνόμαστε για την κατάσταση που υπάρχει. Δεν έχει νόημα. Ε, νομίζω ότι καλό είναι να αναδεικνύονται αυτοί που εξακολουθούν αδιακρίτως να χρησιμοποιούν ε, τα υλικά αυτά κατά του άμαχου πληθυσμού. Ε, είναι μη κυβερνητικοί δράστες, εξεγερθέντες, τρομοκράτες. Πρέπει να πω κύριε Πρόεδρε, ότι προσπαθήσαμε να διαβουλευθούμε ευρέως ε, τον Μάρτιο. Ε, μιλήσαμε για την εκστρατεία κατά των ναρκών, υπάρχει η Γενέβη για την αποναρκοθέτηση, ε, υπάρχει ένα διεθνές ταμείο, το Hello Trust και άλλοι. Επιπροσθέτως έχουμε έγγραφες συνισφορές, από, γραπτές συνεισφορές από άλλους φορείς, από την Υπηρεσία κατά των Ναρκών των Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχει η Ομάδα Δράσης κατά των Ναρκών. Ε, από 14 μέχρι 17 Μαρτίου παραβρεθήκαμε στην 400 η συνεδρίαση του προγράμματος κατά των αρκών στην Γενέβη. Πρέπει να πω ότι εκτιμούμε και σεβόμαστε όλους αυτές τις οργανώσεις και φορείς και τη συμβολή τους. Ωστόσο δεν νομίζω ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να αντανακλά μόνο τις δικές τους απόψεις και τα συμφέροντά τους. Αν θέλουμε να βάλουμε ένα τέλος στην τραγωδία των ναρκών κατά προσωπικού, πρέπει να ληφθούν ορισμένα μέτρα. Και εφιστώ την προσοχή σας ιδίω στην τελευταίο κεφάλαιο της έκθεσης, όπου καλούμε για μεγαλύτερη έμφαση, μεγαλύτερη αξιολόγηση των στόχων, ε, κατάρτιση συνασπισμών σε εκείνες τις χώρες που μπορούν να προσφέρουν περισσότερο είτε σε όρους ανθρώπινου δυναμικού είτε σε όρους ε, χρηματοδότησης. Έκκληση απευθύνεται στην Επιτροπή να δημιουργήσει ένα κονδύλι για την δράση κατά των ε, ναρκών κατά προσωπικού και αυτό έχει συγκεντρώσει τη στήριξη όλων των βουλευτών. Εν κατακλείδη κύριε Πρόεδρε, επαναλαμβάνω την πεποίθησή μας ότι η θέση σε υψηλή προτεραιότητα αυτής της δράσης ε, έχει βελτιώσει την κατάσταση, έχει οδηγήσει σε, καλύτερη υποβολή, καλύτερων εκθέσεων και έχει μειώσει την απειλή κατά της ζωής και της ευημερίας ε, των πληττόμενων πληθυσμών ε, στο χρόνο που μας πέρασε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Πανόρτεν, πρέπει να σας ενημερώσω ότι έχουμε καθυστερήσει λίγο όσο καθυστερήσαμε λίγο με την ψήφιση των προηγούμενων εκθέσεων πάνω στο θέμα του κυρίου Βανόρντεν ε, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και σε άλλες περιπτώσεις. Ο Επίτροπος Φίλε μας περιμένει, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ε, έχουν... Ε, θα ζητήσω λοιπόν αυτοί που ζήτησαν το λόγο να περιορίσουν την παρέμβασή τους σε ένα λεπτό. Κέλλερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Φαν Όρντεν για τη θαυμάσια έκθεσή του. Είναι σημαντική η πρόοδος η οποία επιτεύχθη στον τομέα της αποναρκοθέτησης και του ελέγχου των αρκών ξηρών, ξηράς. Παρ' όλα αυτά, παρά τα θετικά στοιχεία, εξακολουθούν να παραμένουν πολλά προβλήματα, ιδίως σε ανθρώπινο επίπεδο. Ο συνάδελφος Φαν Όρντεν πολύ σωστά αναφέρθηκε στα προγράμματα αποναρκοθέτησης και την αρρωγή που δίδεται στα θύματα των αρκών. Ένα από τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όμως είναι η μείωση των αντιστοίχων προγραμματισμών και την ε, μείωση σε πολυμερή χρηματοδοτικά εργαλεία. <clears throat> Ενώ έχει επιτευχθεί λοιπόν σημαντική και εξαίρετη πρόοδος, εξακολουθούν να παραμένουν μερικές σημαντικές χώρες οι οποίες δεν έχουν προσυπογράψει τη συνθήκη για την απαγόρευση των αρκών Κίνα, Ρωσία, οι Ηνωμένε Πολιτείε μεταξύ άλλων. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η έκθεση είναι μια καλή ευκαιρία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσει πίεση στις χώρες αυτές προς την κατεύθυνση της προσχώρησης στην Σύμβαση της Και αν υπάρχει μονάχα ένας ενεργός χρήστης ο οποίος έχει εντοπιστεί που αυτή τη στιγμή θέτει ακόμα νάρκες στο έδαφος. Υπάρχουν ακόμα σε πολλές χώρες περίπου 30 μη κρατικοί φορείς οι οποίοι προβαίνουν σε ναρκοθέτηση και για τις χώρες οι οποίες δεν έχουν υπογράψει την συνθήκη αυτή για, την, για τις νάρκες έχουν περίπου 160 εκατομμύρια νάρκες που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Ε, Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή που έχει ετοιμάσει ο κ. Βανόργαν αποτελεί πολύ καλή βάση για συζήτηση και αναμένω μια πολύ καλή συνεργασία μαζί του. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να ενισχύσουμε μια πτυχή. Αυτή που έχει να κάνει με την ε, εισφορά των ΗΠΑ και τις προπτικές για το μέλλον. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπογραμμίσουμε το τι κάνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει δεσμευθεί υπέρ του στόχου της απόλυτης εξαφάνισης των αρκών κατά προσωπικό ανατοκόσμου. Πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε την ανθρωπιστική πλευρά του ζητήματος αλλά και τη σύνδεσή του με τις προοπτικές ανάπτυξης που έχουν να κάνουν με ολόκληρες περιοχές και χώρες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το πρόβλημα έχει να κάνει κυρίως με τις πιο φτωχές χώρες στον κόσμο και με την αστάθεια που επικρατεί εκεί. Γι' αυτό και πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει πραγματικά δράση για καταστροφή των αρκών και να υπογραμμίσουμε τις αποστολές μας επιτόπου ώστε να βοηθήσουμε τις προσπάθειες που γίνονται και τοπικά και σε διεθνές επίπεδο για την απενεργοποίηση των αρκών. Δεν έχω περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μου, πάντως θα υποβάλω τροπολογίες για να συμπληρώσω πράγματα τα οποία αναφέρονται ήδη στην, έκφραση, στην έκθεση όσον αφορά την χρήση διεθνών μέσων για την απενεργοποίηση των αρκών. Ευχαριστούμε. Λούνατσεκ, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω κι εγώ να εκφράσω εκ μέρους της ομάδας μου την ικανοποίησή μας για την έκθεση αυτή και για τόσα περιλαμβάνει. Μ' αρέσει και η δομή της έκθεσης όπου αναφέρεται συγκεκριμένες περιπτώσεις. Άρα έτσι έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα για το τι έχει ήδη γίνει και τι μένει να κάνουμε. Θέλω να υπογραμμίσω κυρίως το θέμα της βοήθειας στα θύματα. Μόνο 9% των χρημάτων πάει σε αυτό, μόνο 9% της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ λοιπόν πρέπει να ζητήσουμε περισσότερα χρήματα για την ανακούφιση των θυμάτων, όχι βέβαια σε βάρος της απενεργοποίησης ναρκών. Επίσης πρέπει να κατονομάσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχουν ε, η τυπογράψη, είτε επικυρώσει, είτε μονογράψει την ε, σύμβαση για την απαγόρευση των ναρκών και να πούμε τι γίνεται στη συνέχεια, με παράδειγμα το σχέδιο Καρταχένας. Επίσης αναφερθήκατε τις διάφορες ε, περιπτώσεις μεταξύ των οποίων ε, τα εκρηκτικά που έχουν μείνει από τον πόλεμο ή τις ε, βόμβες κατακαιρματισμού. Είναι και αυτά σημαντικά θέματα. Πολλές φορές έχουμε πολλούς οργανισμούς που δρούν σε ένα και το ίδιο πεδίο. Τώρα δεν ξέρω τι είναι το καλύτερο να κάνουμε για να βοηθήσουμε τις χώρες που έχουν ανάρκειες. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και θα ήταν καλό να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από εσά, από τις ΗΠΑ να μας δώσουν στοιχεία πριν και μετά το 2007 για να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος δρόμος όσον αφορά τις προβλέψεις χρηματοδότησης. Λέζιν, τώρα ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Φανόρντεν και για την επιμονή σας επίσης γιατί αυτό το θέμα ήταν κάτι το οποίο χρειάστηκε και πολλή προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί και εγώ αγωνιστικά για το θέμα αυτό. Είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε λοιπόν όλε τι ψυχές του ζητήματο και η πολιτική μου ομάδα και εγώ χαιρετίζουμε ιδιαίτερα την έκθεση αυτή και με τροπολογίε θα αντιμετωπίσουμε το θέμα τη ε, χρησιμοποίηση των αρκών ε, κατά προσωπικού από μη κρατικέ ε, οντότητες. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και αυτό το θέμα. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στον ε, εισηγητή Βαν Όρτεν για τα τελικά σχόλια πριν να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον Επίτροπο Φίλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τα για νεόδαρα και πολύ χρήσιμα σχόλιά τους. Πολλά από τα θέματα που ε, έθιξαν ε, είναι καθόλου αθεμητά και νόμιμα. Μπορούμε να τα συζητήσουμε και να συνεργαστούμε εξάλλου δεν έχει ολοκληρωθεί η συνεργασία, ε, δεν τόνισα το εξής. Δεν ήθελα να αφιερώσω πολύ χρόνο για να κάνω μια εκτενή παρουσίαση. Είχαμε πολλές εκθέσεις για το θέμα της ε, αποναρκοθέτησης ε, εδώ στο Κοινοβούλιο και έχουμε ξοδέψει πολύ χρόνο να τα συζητάμε και έχω επίγνωση αυτών των συζητήσεων, αλλά στον περιορισμένο χρόνο και χώρο που έχω στη διάθεσή μου, προσπάθησα να δώσω έμφαση στο πώ θα μπορέσει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδο, γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Συμφωνώ με τα σχόλια της κυρίας Λούνατσεκ για τη σημασία τη βοήθεια προ τα θύματα. Ε, ήταν προτεραιότητα, υψηλή προτεραιότητα στο παρελθόν. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από 15 χρόνια ε, διοχέτευσε πολλούς πόρους για τη βοήθεια των θυμάτων. Συστάθηκε το Διεθνές ε, Ταμείο και, μια, και σε συνεργασία με την Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού υπήρξε ειδική συνεργασία από αυτόν για τα πυρομαχικά διασποράς. υπάρχει, ξεχωριστή έκθεση για τα πυρομαχικά διασποράς. Φυσικά όταν αποναρκοθετεί κανείς εκτάσεις αφαιρεί ό,τι υπάρχει, όλα τα εκρηκτικά υπολείμματα του πολέμου. Ε, αλλά εγώ προσπαθώ ε, να να έχω στο επίκεντρο ιδιαίτερα τις νάρκες κατά του προσωπικού. Τώρα για το κονδύλι του προϋπολογισμού. Αυτό δημιουργεί κάποιες διχογνωμίες. Σίγουρα όλοι όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ε, θέλουν πολύ να υπάρχει ένα ενιαίο κονδύλιο ε, τόσο για το ύψος του ποσού όσο και για τη διαφάνεια. Ε, γιατί διαφορετικά είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσουμε και να ελέγξουμε πόσα χρήματα πραγματικά δαπανώνται στα θέματα αυτά, για τα θέματα αυτά. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να το εξετάσουμε. Κύριε Πρόεδρε, κατανοώ ότι δεν έχουμε χρόνο. Ε, αναμένω τα σχόλια και τις προτάσεις των συναδέλφων και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε ίσως και διμερώς να τα συζητήσουμε κάποια από αυτά. Ε, προσβλέπω στην καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βαν Εκτιμώ την τελική σας παρέμβαση, επιδεικνύεται πνεύμα συνεργασίας. Ε, όπως είπα και στην αρχή, θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε και να τα συζητήσουμε πιο εκτενώς. Στη συνέχεια Υπάρχει ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Φίλε για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου των Εξωτερικών Υποθέσεων στις 12 Απριλίου. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Ζητώ λοιπόν να παραμείνουν μόνο οι βουλευτές και οι αρμόδιοι υπάλληλοι. Οι υπόλοιποι παρακαλώ να εγκαταλείψουν την αίθουσα πριν να ξεκινήσει ε, η επόμενη συζήτηση. Θα σταματήσουμε λοιπόν για λίγα λεπτά.